Okay, friends, it's... Uh, Φίλοι μου, είναι 9 και 20. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία. Οι σοσιαλιστές ζήτησαν ονομαστική ψηφοφορία στις προσθήκες από 1 έως 6 στη συνεισφορά της Επιτροπής Απασχόλησης στον διαρθρωμένο διάλογο ή δομημένο διάλογο. Ονομαστική ψηφοφορία. Είναι κανείς κατά. Υπέρ. Ποιος είναι υπέρ της ονομαστικής ψηφοφορίας. Έχουμε πάνω από 11. Άρα θα ξεκινήσει η ψηφοφορία. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προσθήκη 1. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Προσθήκη 2. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται επίσης με τρεις ψήφους περισσότερες, όπως και η προηγούμενη. Προσθήκη 3. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με πέντε ψήφους περισσότερες. Προσθήκη 4. Το ίδιο ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται με 36 ψήφους. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προσθήκη 5. Ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη ψηφοφορίας. Λήξη. Εγκρίνεται με 25 ψήφους. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για την προσθήκη 6. Έναρξη ψηφοφορίας. Λήξη. εγκρίνεται με δύο ψήφου. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι πρέπει να το ελέγξουμε. Ναι, ξεκινάει η ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη συμβιβαστική 10. Πέρασε. 46 υπέρ. Τέλεια. Αλλά μόνο ένας ή δύο είχαν σηκώσει τα χέρια. Ψηφίζουμε τη συνεισφορά της Επιτροπής στον διερθρωμένο διάλογο υπέρ. Ονομαστική ψηφοφορία. Έχει ζητηθεί. Πέρας. Εγκρίνεται με 24 ψήφους υπέρ. Και ευχαριστούμε όλους τους ψηφίσαντες και όσους ενεπλάκησαν στο φάκελο αυτό. Πάμε στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης. Συνθήκες εργασίας και επισφαλής απασχόληση. Ξεκινούμε με τη συμβιβαστική J. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Π υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AK υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 88 όχι καταπίπτει. Και η 391. Καταπίπτουν όλα μέχρι τη σελίδα 3. Πάμε στο 102. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Να το επαληθεύσουμε. Τροπολογία 102. Έναρξη ψηφοφορίας. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 102. Πέρασε. Εγκρίνεται με τρεις ψήφους. 103 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 104. Προφορική τροπολογία που ζήτησαν οι σοσιαλιστές υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το επαληθεύουμε. Την 104 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με δύο ψήφους. 105. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 106. Υπέρ. Απο... Ε, κατά. Αποχές. Θα έλεγα ότι εγκρίνεται. Να το ελέγξουμε, θέλετε, ναι. Την 106 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 28 ψήφους, 107 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα έλεγα ότι εγκρίνεται. Το επαληθεύουμε. Ψηφίζουμε την 107 άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται με τρεις ψήφους. Συμβιβαστική R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. T υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στη σελίδα 7. Συμβιβαστική AM υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AO υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική U υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 163 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 164 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 165 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Επαληθεύουμε την 165 διά της ηλεκτρονικής οδού. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 28 ψήφους. Συμβιβαστική Β, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 178 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική AN υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική W υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 194 υπέρ. Κατά. Αποχές να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Θα έλεγα ότι απορρίπτεται. Όχι. Απορρίπτεται, ναι. 195. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 196 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 197 υπέρ. Κατά. Αποχές. Τη ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 197. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται με 30 ψήφους. 198 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα έλεγα ότι απορρίπτεται. Θέλετε να το ελέγξουμε. Καλώς. Ξεκινάει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται με 27 ψήφους. Συμβιβαστική Y υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Z υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 205 ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 206 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 207 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική AA υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. AB συμβιβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AT υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Σελίδα 13. AS συμβιβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 223 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική AC υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AD υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Σελίδα 14. Συμβιβαστική X υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.39 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 240 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα έλεγα ότι απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 240 ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. Με μεγάλη πλειοψηφία. Συμβαστική ΑΕ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AF υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AG υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AP υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 253. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Τμήμα 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Και θα έλεγα ότι εγκρίνεται. Τμήμα 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα έλεγα ότι εγκρίνεται. Τροπολογία 2.55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 259 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 260 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 262 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ελέγχουμε τη 262. Την επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται κατά τρεις ψήφους. Πάμε τώρα στην 264 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε την 264. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Με μεγάλη πλειοψηφία. Συμβιβαστική AH υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. Γι' αυτό και πάμε στην 2.75 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2.76 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2.54 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Επαληθεύουμε διά της ηλεκτρονικής οδού την 254. Πέρας. Εγκρίνεται με 35 ψήφους. 2.78. Τροπολογία 278. Υπέρ. Καλώς. Την 277. Ποιος είναι υπέρ της 277. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην 278. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 279. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 280 το πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τρίτο, τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 281. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα. Άγκρι 17. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πάμε τώρα στη συμβιβαστική AI. Ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Γι' αυτό και πάμε στην 289. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 290 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.91 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.92 ψηφοφορία κατά τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα της 292. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το πρώτο τμήμα της 292ης τροπολογίας. Πέρας της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και τώρα βλέπουμε ότι απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.93 υπέρ. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Το πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.94. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.95. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AL. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική... Όχι, τροπολογία 301 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται επαληθεύουμε την 301 διά της ηλεκτρονικής οδού, πέρας της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, απορρίπτεται. 302 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική AJ υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 304 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά την 304 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 305 καταπίπτει. Συμβιβαστική AR υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AQ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τη συμβιβαστική AQ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Με μία ψήφο. 3.14 καταπίπτει. 3.15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα έλεγα ότι εγκρίνεται. Το ελέγχουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Όχι, απορρίπτεται. 3.16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.19 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Γι' αυτό και πάμε στη σελίδα 24, η τροπολογία 23 της Άγκρη, υπέρ. Κατά. Πολύ λίγοι σήκωσαν τα χέρια τους. Ψηφίζουμε ξανά την Άγκρη 23, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άγκρη 1, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άγκρη 2, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άγκρη 3, υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 4 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 5 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ναι, εγκρίνεται. Άγκρι 7 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 8 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 9 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 11 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 12 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 13 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 14 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άγρια 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρη 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρη 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρη 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρη 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρη 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η πρώτη της Επιτροπής Γυναικών υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική AB υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΦΑΜ 7 υπέρ κατά αποχές θα έλεγα ότι εγκρίνεται. Η ΦΑΜ 7. Η 8 της Επιτροπής ΦΑΜ. Υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. ΦΑΜ 9. Όχι 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. ΦΑΜ 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται.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 αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 και 9 είναι ταυτόσιμες. Υπέρ. Οι 8 και οι 9 είναι μαζί. Όχι. Υπάρχει λάθος, υπάρχει λάθος στον κατάλογο ψηφοφορία. 8 και 9 μαζί. Συγγνώμη για το λάθος στον κατάλογο. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά αποχές θα έλεγα ότι εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Αποκινούμε την 17. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 15 και 16 ταυτόσημες. από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΦΑΜ, αιτιολογική σκέψη 2, υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 20 και 27 ταυτόσιμες από κοινού υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 22 Επίσης από κοινού με την 23 ταυτόσημες <clears throat> υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται φάμε με τη λογική σκέψη 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική A υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική B υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική E υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική και στη σελίδα 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία συμβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 55 υπέρ κατά αποχές θα έλεγα να επαληθεύσουμε την 55 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται με 8 ψήφους πλειοψηφία. 56 υπέρ κατά αποχές θα έλεγα απορρίπτεται. Να επαληθεύσουμε την τροπολογία 56. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 57 υπέρ κατά αποχές θα έλεγα εγκρίνεται συμβιβαστική G, επαλήθευση της τροπολογίας 57, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας και εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 71 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται επαλήθευση της τροπολογίας 71, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, απορρίπτεται. Φαμ αΐ, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, αγκριντή, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, φαμτί, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται φαμιού υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική N Θέλετε επαλήθευση της τροπολογία 77. Ας την επαληθεύσουμε, την τροπολογία 77. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας εγκρίνεται με 41 ψήφους. Συμβιβαστική εν υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 80 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ΟΟΥ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι J υπέρ κατά αποχές. Πρέπει να την επαληθεύσουμε την agri J. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρας. Εντάξει, πέρας. Απορρίπτεται. Φαμβή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Φαμέι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θα ελέγξουμε την ΦΑΜΕΙ. άρχεται πέρας πληροφορίας εγκρίνεται με 11 ψήφους. Φαμπή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται φανδί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται φαμ ή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται φαμεφ όχι συμβιβαστική αιγιού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται φαμκέι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται φαμ -ο, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, φαμ εσ, υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση της φαμές, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, εγκρίνεται με 23 ψήφους. Φαμ, ποια είναι η επόμενη. Άγκρι A. Υπέρ. Συγγνώμη. Εντάξει. Ψηφίσαμε ξεχωριστά επί της Άγκρι A. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι B υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι C υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αγρι E υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Agri F υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Agri G υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αγρι H υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Agri I υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Agri K υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική AW υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε επί του σχεδίου έκθεσης όπως τροποποιήθηκε η ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται με 38 ψήφους, μία κατά. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή και την ομάδα του. Οπότε προχωρούμε στο σχέδιο γνωμοδότησης για τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκών τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλών δεξιοτήτων. Θα αρχίσουμε με τη συμβαστική τροπολογία 11. Uh, ε, ξεκινούμε ψηφίζοντα ε, ψηφίζοντας ε, την συμβαστική 11 Η κατά εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 6 που είναι προσθήκη στη συμβαστική 12 υπέρ κατά στην δεύτερη σελίδα τροπολογία 6 αποτελεί προσθήκη στην συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πιστεύω Τροπολογία 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 8, 78, 79 και 74 ψηφίζονται από κοινού υπέρ κατά αποχές ας το ελέγξουμε άρχιτη ψηφοφορία λήξη απορρίπτεται 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ελέγχουμε την 79. 75. Διορθώνει πρόεδρος. Λήξη της πληροφορίας. Απορρίπτεται. Με 25 ψήφους. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Οπότε πάμε στην 76, 77 και 78. Κοινή ψηφοφορία. 79 και 80 καταπίπτουν. καταπίπτει η 9, οπότε ψηφίζουμε για την 76, 77 και 78. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 79 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 80 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ελέγχουμε την 80 Έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη. Και απορρίπτεται. 81, 82, 83. Κοινή ψηφοφορία. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 14 συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 11 και 93 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Υπήρξαν αρκετοί που δεν ψήφισαν. Έναρξη λοιπόν της ε, ψηφοφορίας ε, για την τροπολογία 11 και 93, λήξη της ψηφοφορίας και έχει απορριφθεί. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές. Θα την ελέγξουμε. Συμβαστική 2, έναρξη της ψηφοφορίας, λήξη. και εγκρίνεται. Συνεχίζουμε στις ε, συμβιβαστικές 10, 15 και 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές θα έλεγα ότι απορρίπτεται αλλά θα την ελέγξουμε Έναρξη της ψηφοφορίας, λήξη και εγκρίνεται. 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίν, ε, απορρίπτεται. Ελέγχουμε την 17. Έναρξη της ψηφοφορίας για τη 17 λήξη Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Απορρίπτεται λοιπόν. 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 116 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 117 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ή 18 και 118 υπέρ, κατά, αποχές, αν πω εγκρίνεται, αλλά ας το ελέγξουμε. Έναρξη λήξη της ψηφοφορίας. Ναι, εγκρίθηκε με μία ψήφο. 19 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται ελέγχουμε την 19 έναρξη της ψηφοφορίας λήξη ψηφοφορίας και έχει εγκριθεί συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 123 υπέρ κατά απορρίπτεται, εγκρίνεται. Ας ελέγξουμε την 123. Λήψη. Και απορρίπτεται με 37 ψήφους. Η 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 22 και μαζί με την 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 23 μαζί με την 127 και την 128 υπέρ κατά αποχές θα το ελέγξουμε έναρξη ψηφοφορίας λήξη και απορρίπτεται συνεχίζουμε στην 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 130 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, πάμε τώρα στις αιτιολογικές σκέψεις. 6. Η τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε την τροπολογία 27 έναρξη της ψηφοφορίας λήξη ψηφοφορίας και απορρίπτεται με 23 ψήφους 28 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε και την 28. Έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη. Και απορρίπτεται με 25 ψήφους. Πάμε στη συμβεβαστική 6. Υπέρ, κατά, αποχές συγκρίνεται Τροπολογία 38 μαζί με την 39, 40 και 41 υπέρ κατά αποχές θα έλεγα ότι απορρίφθηκε, αλλά θα την ελέγξουμε. Έναρξη. Λήξη της ψηφοφορίας. Και έχει απορριφθεί με 24 ψηφούς. 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αιτιολογική σκέψη. Τροπολογίες 43, 44, 45, 46 από κοινού. Υπέρ, κατά, αποχές. Θα το ελέγξουμε. Έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη. Και έχει απορριφθεί. 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 και 49 από κοινού υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται θα ελέγξουμε όμως ε, την συμβιβαστική 1 λήξη της ψηφοφορίας και εγκρίνεται με 24 ψήφους και η τροπολογία 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και ε, τώρα ε, ψηφοφορία επί του συνόλου ε, του κειμένου όπως έχει τροπολογηθεί έναρξη της ψηφοφορίας λήξη. Σας ευχαριστώ ε, προς ε, τους εισηγητές, τον εισηγητή, έχει κληθεί. Yes. You know, we are now... Και ε, τώρα θα ε, μεταβούμε στην αίθουσα PHS 3C50 ε, ε, για μια συνεδρίαση και στη συνέχεια θα επιστρέψουμε εδώ. Το ε, θέμα μετά από την ακρόαση που έχουμε τώρα είναι το τι ε, θα συμβεί με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ε, και τον οριστέντα διευθυντή, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας. Τώρα για μια μισή ώρα λοιπόν θα πάμε στην αίθουσα PHS 3C 50 ε, για μια ε, συνάντηση με την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και στη συνέχεια στις 11 και 45 θα πρέπει να είμαστε και πάλι εδώ ε, για να ενημερωθούμε σχετικά με το τι έγινε με τον οριστέντα διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.